Δημοκρατίας, κύριε Σεψή, κυρία Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρία Μογκερίνη, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε όλοι αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε την υψηλή τιμή να υποδεχόμεθα σήμερα τον Πρόεδρο της Τινησιακής Δημοκρατίας. Είμαι συγκινημένος από την παρουσία σας εδώ κύριε Πρόεδρε ένα χρόνο μετά από την τελευταία συνάντησή μας στην Τινησία. Θέλω λοιπόν εκ νέου να σας ευχαριστήσω για την θερμοτάτη φιλοξενία της χώρας σας. Στην αρχή της παρουσίας σας εδώ, έστω και με λίγη καθυστέρηση, να σας συγχαρώ. Ε, γεννηθήκατε στις 29 Νοεμβρίου του 1926 δεν λέμε 90 χρόνια, λέμε 9 και μετά βάζουμε το 0. Χρόνια πολλά. Έτσι μου είπε να πω λοιπόν ο πρόεδρος, γι' αυτό και εγώ λέω 9.0. Κύριε Πρόεδρε, εδώ είστε ανάμεσα σε φίλους. Εδώ είστε ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι πιστεύουν στο δημοκρατικό μέλλον της χώρας σας. Μέσα σε πέντε χρόνια η πορεία της χώρας σας ήταν μια πορεία έκτακτη, εξαιρετική. Η χώρα σας σήμερα θεωρείται πρότυπο ανοχής, θεωρείται πρότυπο πλουραλισμού Μέσω του συντάγματος δίδονται εγγυήσει για το κράτος δικαίου και την ισότητα και τις ελευθερίες όλων. Σε μια εποχή όπου όλοι οι λαϊκιστές ε, ανεμίζουν τον φόβο, το μήνυμα που στέλνει η δική σας χώρα είναι πολύτιμο. Κατά τη διάρκεια της, ε, πολι... της ε, επίσκεψής μου της επίσημης στην Τινησία και στο Σούσι, καταφέραμε να διαπιστώσουμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η χώρα σας σε καθημερινή βάση. Πάντως πιστεύω ότι η χώρα σας παρά τις δυσκολίες της έχει μια, ένα τεράστιο πλούτο, τα νιάτα της, τα δημιουργικά και δραστήρια νιάτα που είναι έτοιμα να δώσουν αγώνα για το μέλλον και την ευημερία της χώρας. Αυτό είναι ένα τρομερό πλεονέκτημα το οποίο σας χαρακτηρίζει. Θα γίνουν οι απαιτούμενε μεταρρυθμίσεις έτσι ώστε να ενθαρρυνθούν και οι τοπικοί επενδυτές και οι εταίροι εκτός χώρας όπως το απέδειξε χθε και η συνάντηση των επενδυτών για την χώρα σας. Η Τινησία δεν είναι μόνη. Η διάσκεψη που έγινε στην αρχή της εβδομάδας για τις επενδύσεις στην Τίνιδα αποδεικνύει ακριβώς το ενδιαφέρον του διεθνούς οικονομικού παράγοντα. Συνεπώς λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τιμήσει τις υποχρεώσεις τις οποίες έχει αναλάβει. Γιορτάζουμε φέτος 40 χρόνια διμερούς συνεργασίας που έχει καταστήσει την Ευρώπη τον πρώτο εμπορικό σας εταίρο και είναι κάτι το οποίο μας κάνει υπερήφανος αποφασίσαμε να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Αναλάβαμε την υποχρέωση να δημιουργήσουμε μαζί σας μια εταιρική σχέση ενισχυμένη και να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε σε πάρα πολλούς τομείς γιατί οι σχέσεις μας έχουν φτάσει σε έναν θα έλεγα στρατηγικό, έχουν αποκτήσει ένα στρατηγικό χαρακτήρα ο οποίος δεν μπορεί πια να αλλάξει. Έχουμε ένα κοινό όραμα για το μέλλον πρόεδρε οι νέοι και από τις δύο πλευρές της Μεσογειακής Λεκάνης συμμερίζονται τις ίδιες ε, προσδοκίες, θέλουν να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα, να ταξιδεύουν, να σπουδάζουν και να εργάζονται. Και πρέπει λοιπόν και εμείς να ανταποκριθούμε στις θεμητές τους προσδοκίες. Γι' αυτό ακριβώς και η νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έναν χώρο νεότητας είναι κάτι που αποδεικνύει ότι θέλουμε να υποστηρίξουμε το ταλέντο, θέλουμε να υποστηρίξουμε τον δυναμισμό της νεολαίας της χώρας σας. Αυτή είναι η καλύτερη επένδυση την οποία μπορούμε να κάνουμε προς όφελος του συνόλου της τινησιακής κοινωνίας. Δεν θα πρέπει να αφήνουμε τους νέους να στρέφονται στις δολοφονικές ε, ιδεολειπτικές ε, απόψεις. Πρέπει εμείς να αποτρέψουμε τα μαύρα σενάρια των εξτρεμιστών. Πρέπει εμείς μαζί να αποδείξουμε ότι οι καθολικές αξίες συνδυάζονται με τον ίδιο τρόπο και στην Τινησία και στην Ευρώπη. Γι' αυτό να χαιρετήσω και την πρωτοβουλία την οποία πήρατε ξεκινώντας ε, με την δήλωση της Τινησίας ε, υπέρ της ανοχής και κατά της τρομοκρατίας στο περίφημο μουσείο του Μπάρντο. Να σας διαβεβαιώσω ότι θα είμαστε πιστοί σας σύμμαχοι, θα είμαστε πιστοί σύμμαχοι της νεότητάς σας και των αρχών της χώρας σας. Σας ευχαριστώ για μία ακόμη φορά λοιπόν Πρόεδρε που μας κάνετε την τιμή να είστε ανάμεσά μας σήμερα. Σας δίδω το λόγο.